Καλημέρα σας όλοι, αγαπητοί συνάδελφοι. Ζητά το λόγο ο κύριος Καρίμ ε, και του δίνω το λόγο. Κύριε Καρίμ, έχετε το λόγο. Mr. President, in July last year, Per cortesia, ascoltiamo l'onorevole Karim. Σας παρακαλώ, ας ακούσουμε τον συνάδελφο Καρίν. Προτσέιντα. Σας παρακαλώ, κύριε Καρίν. Το μικρόφωνο λειτουργεί μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Πέρσι τον Ιούλιο περικυκλώθηκε το σπίτι μου στο Ηνωμένο Βασίλειο από ένα όχλο γεμάτο ρατσιστικό και θρησκευτικό ε, μίσος με ε, βίες προθέσεις. Η σύζυγός μου και το παιδί μου ε, κατατρόμαξαν. Δώδεκα ε, πρόσωπα καταδικάστηκαν σε ποινικό δικαστήριο για τις πράξεις αυτές και τα δικήματα. Θέλω να ευχαριστήσω τον πρώην πρόεδρο κύριο Μπούζεκ που καταδίκασε κατά τη θητεία του ε, αυτά τα φαινόμενα και τη συνάδελφο Εμινέ Μποσκούρτ καθώς επίσης και τη συντριπτική πλειονότητα ε, του Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ και την αστυνομία του Λάγκασερ που με βοήθησε και προστάτευσε την οικογένειά μου και με επέτρεψε να συνεχίσω τα κοινοβουλευτικά μου ε, καθήκοντα και τη δικαιοσύνη του Ηνωμένου Βασιλείου που τους προσήγαγε. Σήμερα δεν έχω απάντηση για την 9 χρονικό μου που εξακολουθεί να με ρωτάει γιατί. Εδώ όμως μέσα συμμετέχει ένας ευρωβουλευτής που τότε ε, έδωσε ε, αμέριστη υποστήριξη και βοήθεια σε αυτούς τους ρατσιστές. Και να είστε βέβαιοι ε, για το εξής. Δεν πρόκειται να δηλιάσουμε απέναντι στη δική σας δειλή προσέγγιση. Θα είμαστε ενωμένοι και θα σας αντιμετωπίσουμε. Σήμερα ομιλώ όχι μόνο εξ ονόματος του Κοινοβουλίου, αλλά εξ ονόματος κάθε εχέφρονο πολίτη της χώρας μου και της Ευρώπης. Ευχαριστώ. Πρέγω. Μαν... Prego, parli per cortesia. Παρακαλώ μιλήστε, σας δίνω το λόγο. Η κατάσταση στην Ουκρανία είναι αυτό που θέλω να αναφέρω. Η κατάσταση της πρώην Πρωθυπουργού κυρίας Τιμοσέγκο και προτινόμενο μποϊκοτάρισμα ε, του ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος Ευρώ 2012. Ε, θέλω να το συζητήσουμε στην επόμενη Ολομέλεια του Στρασβούργου κατά τη διάρκεια της συζήτησης για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Ουκρανία. Επίσης θα ήθελα να σας απευθύνω έκκληση να απορρίψουμε το μποϊκοτάζ. Αυτό που θέλουμε εμείς είναι να προωθήσουμε τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Ουκρανία. Οι πάντες, συμπεραμβανωμένες και της αντιπολίτευσης, θέλουν να διεξαχθεί ε, το ε, Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Προδοσφαίρου Ποδόσφαιρο είναι ε, το σύμβολο της υποστήριξής μας. Και σας προσφέρουμε αυτή την μπάλα ως σύμβολο της υποστήριξής μας ε, προς την κυρία Τιμοσέγκο. Και εγώ παίζω ποδόσφαιρο, λέει ο πρόεδρος. Αγαπητοί συνάδελφοι, ξεκινά η ψηφοφορία η οποία θα είναι μακριά και θέλω να εκφράσω την αλληλεγγύη όλη της αιθούση τον κύριο Καδίμα και την προσωπική μου και εν ονόματι του Πρόεδρου Σούλτς. Θέλω να σας πω ότι η γραπτή δήλωση των συναδέλφων Αλμπερτή, Νικολάνσκα, Μπερβίσκα, Ρινάλντι και Σασόλη σχετικά με τη στήριξη